Ladies and gentlemen, Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην ε, τελική συνεδρίαση της Ουκρανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Χαίρομαι που είναι παρόν και ο κύριος Γκρόισμαν που θα, κάνει, θα απευθύνει χαιρετισμό στο κλείσιμο της ε, συνεδρίας και εγώ στη, κατά Λυπούμε που δεν μπόρεσα να έρθω ε, χθες στις εργασίες της πλήρης. Ε, χρειάστηκε όμως ε, για λόγους πένθους οικογενειακού να μεταβώ στην ε, Ιρλανδία. Επέστρεψα όμως και σήμερα είμαι εδώ κοντά σας. Πολλά πράγματα μαθαίνουμε από κάθε μια από αυτές τις συζητήσεις, τις συναντήσεις και βεβαίως περιμένω να ενημερωθώ και πλήρως ε, από τους συνεργάτες μου για τα όσα δημιουργήσαν κατά την απουσία μου. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία αναλογισμού, αφούγκρασης, αφούγκρασμού, συζήτησης και διατύπωση συστάσεων πλέον. Για να αποδώσουμε λοιπόν την πλήρη τους αξία σε αυτές τις προσπάθειες θα πρέπει να συμβούν τα εξής πρώτο και σημαντικότερο, όλοι οι φίλοι και συνάδελφοι από την Ουκρανία να αναλάβουν, να πάρουν στα χέρια τους τη διαδικασία και να αποδηθούν σε αυτήν την προσπάθεια μόνοι τους. Δεν μπορεί να τους επιβληθεί από κανέναν απ' έξω δηλαδή. Τίποτε. Πρέπει μόνοι τους να ενθενιστούν αυτόν τον αγώνα και το πνεύμα το οποίο αναπτύχθηκε εδώ να το διαφυλάξουν μέχρι και το Κίεβο και να το κάνουν να προχωρήσει. Δεύτερο στοιχείο, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζουν τη σημασία της προσπάθειας αυτής θα πρέπει να ξαναφορτίσουν τις μπαταρίες τους και να σας στηρίξουν στην προσπάθεια αυτή για τη μεταμόρφωση, για την βελτίωση της κατάστασης και γι' αυτό με ενδιαφέρον περιμένω να ακούσω τις δύο πρόπτικες από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κύριο Πλένκοβιτς εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλος πυλώνας του εγχειρήματος όχι επιβολητικό τόσο, αλλά διοικητικό. θα είναι οι συστάσει το σημαντικό αυτό κομμάτι των συστάσεων. Και με χαρά βλέπα τον κύριο Σλουζίνσκι από την πλατφόρμα. Και αργότερα περιμένουμε να δούμε και τον κύριο Βέλε, Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να το επιτρέψουν τα καθήκοντά του. Αξιωματούχοι και οι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα υπογράψουν συμφωνία για την ανάπτυξη διοικητικού δυναμικού. Με μια πρώτη συμφωνία, ιστορική πρώτη, που υπογράφεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εν τέλει, και απευθύνομαι σε ένα ευρύτερο ακροατήριο συμμετεχόντων που είναι εδώ παρόντες ε, σήμερα, όλοι οι διεθνείς εταίροι, κράτη, εθνικά κοινοβούλια, μη κυβερνητικέ οργανώσει, άλλα θεσμικά όργανα και ιδρύματα που μπορούν να εμπλακούν θα πρέπει να προσφέρουν τις γνώσεις και την υποστήριξή τους στο Κοινοβούλιο της ε, Ουκρανίας και να βοηθήσουν στην κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων που εσείς θα αποφασίσετε να προωθήσετε στην Ουκρανία. Γιατί η μεταμόρφωση αυτή δεν θα είναι ούτε ευχερής ούτε δωρεάν. Θα χρειαστεί η υποστήριξη όλων των εταίρων κατά τρόπο συντονισμένο, κατά τρόπο εστιασμένο, ώστε να μην γίνεται διπλή προσπάθεια, να μην εκδηλώνεται, να μην αφιερώνονται διπλή πόροι, αλλά οτιδήποτε υπάρχει σαν προσπάθεια, σαν ε, υποστήριξη, σαν καλή θέληση και σαν πόροι να τίνουν συνδυασμένα προς την ίδια κατεύθυνση. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τις οικές μου τοποθετήσεις, θα ήθελα να ακούσω τις πολύ σημαντικέ ε, θέσεις και προοπτικές των δύο κύριων φορέων και δίνω το λόγο στη Helga Schmidt αναπληρώτρια Γενική, Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ψητερικής Δράσης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ και καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της εβδομάδας ε, της Ουκρανίας που πιστεύουμε ότι ενίσχυσε την κοινοβουλευτική διάσταση των σχέσεων ανάμεσα στην Ένωση και την Ουκρανία. Ε, ήταν ε, εντυπωσιακέ οι ε, ομιλίε και πολλέ επαφέ έγιναν στα περιθώρια των ε, επίσημων συνεδριάσεων. Αυτό βοήθησε στο να δημιουργηθούν κοινέ βάσει, ε, πλατφόρμε, ώστε η Ένωση με την Ουκρανία να συνεχίσουν να ενισχύουν του δεσμού του. Αυτό δίνει όχι μόνο βάθος και δυναμική στην κοινή μας ημερήσια διάταξη, αλλά δημιουργεί και σχέσεις και επαφές ανάμεσα στους πολίτες, μα. μας. Συζητήσαμε αυτήν την εβδομάδα τη δικαστική μεταρρύθμιση, την καταπολέμηση διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του διοικητικού τομέα, την αποκέντρωση και πολλά ακόμα. Και Όπω ακριβώ είπε και ο πρόεδρο Κόξε, η Ουκρανία θα πρέπει να αποφασίσει η ίδια πώ θα προχωρήσει σε όλα αυτά. Οι Ουκρανοί οφείλουν να αναλάβουν ε, τα ενία, να... αυτό πιστεύουμε κι εμείς, ε, γιατί τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις είναι πολύ ζωτική σημασία για την αποτελεσματική και βιώσιμη δημοκρατική μεταρρύθμιση. Γνωρίζουμε ότι η μεταρρύθμιση των θεσμών στο πλαίσιο της δημοκρατικής μετάβασης είναι εξαιρετικά περίπλοκο εγχείρημα ως προς αυτό η έκθεση στο νοδικό χάρτη που εσείς ε, υποβάλλατε κύριε Πρόεδρε μετά από την αποδοχή της στην ΕΡΑΝΤΑ, το ευθερίδι αυτό. Ε, θα είναι μια σημαντική συμβολή στην ε, στήριξη των μεταρρυθμίσεων στην ΕΡΑΝΤΑ αλλά και στην Ουκρανία Επίσης, είμαστε, θα δούμε πολύ προσεκτικά αυτές τις συστάσεις για να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε καλύτερα την Ουκρανία να προχωρήσει. Όπως ε, αποδείχθηκε και φάνηκε από την ίδια την διεξαγωγή της εβδομάδας της Ουκρανίας εντό του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου, η Ουκρανία είναι ε, τέρος κλειδί την ε, ε, πολιτική γειτονία και την ανατολική εταιρική σχέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε την ανατολική εταιρική σχέση που είναι το ευρύτερο πλαίσιο σχέσεων με την Ουκρανία μόλις πέρσι. Η διαφοροποίηση και η βελτιωμένη ε, ανάληψη των ε, έργων, των μεταρρυθμίσεων από τους Ουκρανούς θα είναι στη καρδιά της προσπάθειας. Καλωσορίζουμε τη συμβολή της Ουκρανίας στην διαβούλευση και προσβλέπουμε σε περαιτέρω συζητήσεις για την εφαρμογή μετά από τις προτάσεις. Η, πρόσθεση, η προσέγγιση μας στην Ανατολική ε, εταιρική σχέση θα εστιάσει σε πιο στοχοθετημένη ατζέντα συνεργασία και στο να οικοδομήσει την αντοχή του εταίρου μα. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη διμερή συνεργασία, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να διατηρηθεί η ε, γενικευμένη φύση της ανατολικής εταιρικής σχέσης και η πολυμερή συνεργασία που περιλαμβάνει τους έξι εταίρους. Πρέπει να έχουμε αποτελέσματα, θέλουμε δηλαδή στένος και δέσμευση από όλες τις πλευρές για να προχωρήσουμε. Ε, θέλουμε να προωθήσουμε ε, την ε, πέρβαση των τρεχουσών εγχωρίων δυσκολιών ώστε να συνεχίσει η Ουκρανία την πρόοδο που έχει επιτύχει στους τελευταίους 14 μήνες. Τα πολιτικά παιχνίδια δεν θα πρέπει να υπερισχύσουν, να κυριαρχήσουν τις ευρύτερη πρόοδου και πιστεύω ως προς αυτό οι συναντήσεις που είχαμε το δείπνο στο οποίο κάποιοι από εμάς συμμετείχαμε χτες το βράδυ ήταν πολύ σημαντική συμβολή. Μην ε, ε, απογοητευτείτε τώρα, μην τα παρατήσετε. Ο ρόλος της Ράντα ε, είναι σημαντικός για να είναι η κάθε κυβέρνηση υπόλογη και για να ε, περνούν οι απαραίτητοι νόμοι που είναι η βάση για την μεταρρύθμιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπηρεσία δράσης, ε, είπατε εκπρόσωπος, είναι απόλυτα προσιλωμένη στην παρακολούθηση της, Ευρωπα... της Ουκρανίας και έχουμε φορτώσει τις μπαταρίες μας ως προς αυτό κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν τα μέσα υπό την ε, πολιτική γειτονία έχουμε τη Συμφωνία ε, Σύνδεσης και την Εμπορική Συμφωνία που την έχουν διαπραγματευτεί διαδοχικά σε ουκρανικές κυβερνήσεις τώρα είναι ε, στην προσωρινή εφαρμογή ε, εκκρεμεί η πλήρη της, της εφαρμογή και πρέπει η Ουκρανία να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Είμαστε σχεδόν στο τέλος του δρόμου όσον αφορά την απελευθέρωση, την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό νομίζω. Όλοι μας το είπατε τη διάρκεια αυτή τη εβδομάδα. Η πρόοδο που έχει κάνει η Ουκρανία και οι δεσμεύσει τη Ουκρανική ηγεσία να αντιμετωπίσει λίγα ε, προβληματάκια διαφθορά μέσα στο 2016 θα επιτρέψουν στην Κομισιόν να υποβάλει θετική έκθεση το Δεκέμβριο. Η Κομισιόν προετοιμάζει την σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Αλλά θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι δεσμευμένη για να στηρίξει την Ουκρανία στον τομέα της ασφάλειας. Έχουμε μια ευρωπαϊκή υποστολή επιτόπου με ενημερωμένη εντολή που παρέχει στρατηγικές ε, συμβουλές και στήριξη στον ε, μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στην Ουκρανία. Όπως σας είπα, συνεχίζουμε τη γενική στήριξη, αλλά δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την πολιτική βούληση ώστε να γίνουν οι αλλαγές που θέλουν οι ε, οι πολίτες της χώρας αλλά ε, μπορούμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα. η ανατολική εταιρική σχέση ίσως να μην έχει προχωρήσει αρκετά σε σχέση με τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας. Όμως θα πρέπει να σας πω ότι η Συμφωνία Σύνδεσης μαζί με την Εμπορική Συμφωνία μας δίνει την, ευκαιρία, δίνει την ευκαιρία στην Ουκρανία να γίνει μια πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα με πλήρως λειτουργούσα δημόσια διοίκηση, ε, οικονομία της ε, αγοράς και πραγματικά δημοκρατικούς θεσμούς. Για το πρόγραμμα απελευθέρωσης των θεωρήσεων θα επιτρέψουμε σε σύντομα στους Ουκρανούς να μπορούν να επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να χρειάζεται να πάρουν βίζα. Ε, αυτό νομίζω θα αυξήσει την αίσθηση της ε, συντροφικότητας. Ε, κάτι που παρατήρησε κάποιος συνδετημόνας στο χτωσινό δείπνο. Βέβαια, Υπάρχουν οι δυσκολίες ε, στις σχέσεις με τη Ρωσία, ιδιαίτερα όσον αφορά την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας και της Σεβαστούπολης και τη συνεχιζόμενη ε, σύγκρουση προς Ανατολάς. Εμείς ε, είπαμε ότι δεν μπορούν να επανέλθουν στη συνηθισμένη τους κατάσταση σχέση μεταξύ Ένωσης και Ρωσίας μέχρι ώστε να βρεθεί μια λύση σε αυτή την κρίση. Αν δείτε τα περιοριστικά μέτρα για τη Ρωσία και τη συνεχιζόμενη στήριξή μας για την Ουκρανία και άλλους γείτονες, έχουμε αποδείξει πόσο αποφασισμένοι είμαστε σε αυτό το τομέα. Οι συμφωνίες του ΜΙΣΚ θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως ε, αυτό συμπεριλαμβάνει την απόσυρση όλων των ξένων ε, στρατιωτικών ε, μονάδων καθώς και την τον ουκρανικό έλεγχο των συνόρων. Αλλά θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι όλες οι πλευρές θα πρέπει να δεσμευτούν για πλήρη εφαρμογή. Ξέρω πως είναι δύσκολο να συνεχίσει κανείς στην πολιτική αυτή γραμμή και να κάνει συμβιβασμού όταν ξεκολουθούν οι παραβιάσεις της ανακοχής. Όμως η συμφωνία του Μίνσκ ε, ε, προβλέπει την κυριαρχία στις ε, περιοχές το Λένς και το Χατ. Αυτό σημαίνει πως η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερα από τη δική της πλευρά. Έχει ήδη καταβάλει προσπάθειες για να λειτουργήσει η ειρηνική λύση. Γνωρίζουμε τα αίτια της σύραξης, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, καταλαβαίνουμε τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ε, Ουκρανία και αυτό το υπογραμμίζω και προσωπικά σε κάθε διάλογο που έχω με τρίτες χώρες διότι κάποιες φορές δεν γίνεται πλήρως αντιληπτό εκτός της Ένωσης αλλά θα ξαναπώ ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει υπευθυνότητα και να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Πάντως θα πρέπει να δούμε ότι μετά από δύο χρόνια η επιδεινούμενη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Χερσόνησο προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι η Ένωση δεν αναγνωρίζει την παράνομη προσάρτηση της περιοχής και θα συνεχίσει να εφαρμόζει αυτή την πολιτική μη αναγνώρισης. Γνωρίζω πως τα μέλη του Κοινοβουλίου και της Ράντα θα συνεδριάσουν σύντομα και πάλι για την ε, πέμπτη τακτική ε, συνεδρίαση, κοινοβουλευτική συνεδρίαση της Euronest, την κοινοβουλευτική πτυχή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και ότι θα είναι μια ακόμα ευκαιρία για να συζητήσουμε το ρόλο των κοινοβουλευτικών ανταλλαγών και συνεργασίας. Ε, η έμφαση του Ευρωκοινοβουλίου για την Ουκρανία και ενισχυμένη σχέση με την Ράντα είναι ένα παράδειγμα των στενών και βαθιών σχέσεων. Η ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική για να επιτύχει η χώρα και όλοι θέλουμε να επιτύχει η χώρα. Γι' αυτό και ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες σας και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Thank Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμβολή σας στη συζήτηση. Κάνατε μια γενική επισκόπηση της κατάστασης. Για αυτή την μεταρρυθμιστική διαδικασία στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας με ενθαρρύνει η δέσμευση που έχετε αναλάβει για να μας υποστηρίξετε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό. Και η παροχή συμβουλών, γιατί για συμβουλές πρέπει δεν πρόκειται εμείς να αποφασίσουμε τι συμβαίνει στην εσωτερική τάξη της Ουκρανίας. Η παροχή συμβουλών λοιπόν είναι ε, σημαντικό τμήμα της διαδικασίας. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Σέμιρακ. Δεν είστε στο οπτικό μου πεδίο και σας ξέχασα. Θα σας δώσω το λόγο εν το χρόνο. Θα δώσω όμως το λόγο προς το παρόν στον Αντρέη Πλένκοβιτς που είναι συμπρόεδρος ε, της ε, αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, Επιτροπή Σύνδεση, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ Ουκρανίας. Θα ήθελα τώρα που έχουμε περάσει στη φάση της έκθεσης για την εξολόγηση των αναγκών να μας δώσετε μια συγκεκριμένη άποψη από πλευράς του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε Πρόεδρε. Ε, κύριε Σπίτ, Πρόεδρε του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, ε, κύριε Σμίτ, σας ευχαριστούμε που μιλήσατε για τις προκλήσεις ως προς την ασφάλεια θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί στα πλαίσια της άτυπης Επιτροπής Σύνδεσης, αγαπητά μέλη του Ουκρανικού Κοινοβουλίου, αγαπητοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Σίβιτς, κύριε Κόβαλ, η προκάτοχή μου. Θα ήθελα για την τρίτη συναυτή ημέρα ε, να τονίσω πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, Ουκρανία, για την ε, πολιτική χειραφέτηση αυτή της χώρας, τη σημασία που έχει αυτή η χειραφέτηση για τις αξίες σε παγκόσμιο επίπεδο, για την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως για την αλληλεγγύη που δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς μια χώρα που έκδηλα έχει ε, προκρίνει πλέον αυτή την άγουσα, δηλαδή το δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά εχθές στους διαλόγους υψηλού επίπεδου είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε εμπειρίες ε, και ιδέες ε, με τα, τους ειδικού από την κοινωνία των πολιτών και τα μέλη του Ουκρανικού Κοινοβουλίου. Ήταν ιδιαίτερα γόνιμο το έδαφος ε, για τις συζητήσεις. Ε, πέρα από τους βουλευτές του Ουκρανικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε ανταλλαγή ανάμεσα και στους, στα μέλη του ίδιου του Ουκρανικού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα καρποφόροι συζητήσεις που κάναμε. Στο Κοινοβούλιο, καλύτερη πρακτική που έχουμε γιατί μιλάμε για το εθνικό ή το ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αυτή η ανταλλαγή απόψεων και αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε ως μήνυμα και νομίζω ότι το είδατε μας τις τελευταίες δύο ημέρες. Με αυτήν την εβδομάδα για την Ουκρανία, για την Ουκρανία και το πρόγραμμα που ε, ήταν ιδιαίτερα επίμουθο στη σύνταξή του με απασχόλησε τους τελευταίους μήνες και όχι μόνο εμένα αλλά και τους συναδέλφους μου και ακολουθεί <laughs> λοιπόν αυτή την εβδομάδα μία έκθεση αξιολόγηση των αναγκών όπως είπε είπε ο πρόεδρος Πατ και θα συμπεριλάβουμε όλες τις συμβουλές από όλους τους συνομιλητές μας χάρη στις οποίες έχουμε εντοπίσει και προσδιορίσει 52 συστάσεις και πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά σας σε αυτήν την διαδικασία διότι αυτή η άσκηση που γίνεται δεν αφορά μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κηρύττει τι πρέπει να γίνει ή οποιοδήποτε άλλος που θα προσπαθούσε να κηρύξει και να μας πει ε, πώς θα πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον στην Ουκρανία. Όχι, έχουμε συλλέξει στοιχεία και ερμηνεύσει σημάδια ούτω ώστε να μεταρρυθμιστεί το κοινοβούλιο ε, και να γίνει δίτικο στραφές, να εξυγχρονιστεί το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ε, και νομίζω ότι αυτό είναι ε, το βασικό μήνυμα σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την Ουκρανία και που αναλαμβάνουμε εδώ στο κοινοβούλιο. Κάτι που έχει κέρια σημασία είναι πως οι συστάσεις που έχουμε δεν είναι μόνο άσκηση επιχάρτου, συνδέονται από την ετοιμότητα, τη βούλη θέληση του Κοινοβουλίου να ε, χορηγήσει τα απαιτούμενα κονδύλια για να διευκολύνει την εφαρμογή των συστάσεων. Αυτό είναι σημαντικό. Κάθε φορά που συστήνουμε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία τα πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει σε συγκεκριμένο οδικό χάρτη, θα υπάρξουν ε, κονδύλια ε, στην, στη, στο, στη διεύθυνση για την υποστήριξη του εκδημοκρατισμού που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά, θα εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι την, ε, το πέρας της τωρινής θητείας. Το Κοινοβουλίο. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Χρειαζόμαστε χρόνο για να υλοποιήσουμε αυτήν την εταιρική σχέση και να γίνει αυτή η αδελφοποίηση, ας το πω έτσι, περί αυτού πρόκειται ανάμεσα στα δύο κοινοβούλια ο ε, πρόεδρε της Βουλής, ε, κύριε Γκρόισμεν, ε, ε, αγαπητοί βουλευτές του Ουκρανικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, ε, χωρίς τη δική σας βοήθεια είναι αδύνατο να φέρουμε σε πέρα σε αυτό το τεράστιο εγχείρημα. Μιλάμε για την αρχή περισσότερα για περισσότερα όταν μιλάμε για την πολιτική ή και ανατολική γειτονία. More for more. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε το πρόγραμμα ανάπτυξη ενδογενών ικανοτήτων, capacity building και αυτό χρειαζόμαστε αλλά με ευέλικτο τρόπο. Θα ήθελα να σχολιάσω τις συγκεκριμένες συστάσεις από τα διάφορα πάνελ υψηλού επίπεδου. Ε, σχέσεις ανάμεσα στην εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία. Πολύ χρήσιμες εργασίες αυτού του πάνελ. Και ε, είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε και με τον ε, μεγάλο φίλο της Ουκρανίας, τον πρώην πρόεδρο Μπούζεκ και εδώ εντοπίσαμε διάφορες διαστάσεις του θέματος ε, να δούμε πώς ε, ο ενισχυμένος συντονισμός ε, του νομοθετικού και του εκτελεστικού έργου μπορεί να επιτευχθεί. Μία διοργανική συμφωνία, παραδείγματος χάρη, ανάμεσα, για τη συνεργασία ανάμεσα στο Ράντα, στο Κοινοβούλιο και το Κυβερνητικό Επιτελείο. Η εμπειρία που έχουμε εδώ από τη συνεργασία Κοινοβουλίου και Επιτροπής μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα σύστημα κοινών ελέγχων που θα μας οδηγήσει ε, προς τα μπροστά. Κατά τα λοιπά θα χρειαστούμε τις καλύτερες ε, πρακτικές ε, των συναδέλφων για την νομοτεχνική, νομοπαρασκευαστική διαδικασία ε, ποια είναι η πρόθεση, ο σκοπός, το σκοπούμενο κάποιου νομοθετήματος πέρα από την πολιτική φιλοδοξία σε κάθε μία από τις φάσεις της υλοποίηση ε, θα πρέπει να υπάρχει συνειδητοποίηση και γι' αυτό μπορείτε να συντάξετε πράσινες βίβλους, ε, λευκές βίβλους, ανακοινώσεις ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς επαρκώς νωρίς να εμπλέκονται, να συμμετέχουν στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία και μαζί με την αξιολόγηση, τη μελέτη αντικτύπου, να έχουμε μια πλήρη εικόνα σε σχέση με το τι σημαίνει να υιοθετηθεί ένα νομοθέτημα και ποιε επιπτώσει θα έχει η εφαρμογή του για την κοινωνία, αλλά και ποιε οικονομικέ επιπτώσει θα έχει. Επίση, τι άλλο μπορούμε να βοηθήσουμε εμεί από πλευρά του Κοινοβουλίου. Ενίσχυση του ρόλου των επιμέρου επιτροπών του Κοινοβουλίου και για την νομοθετική διαδικασία, αλλά και για την εποπτεία του ε, ε, κυβερνητικού έργου. Άτυπο δίκτυο, παραδείγματο χάρη ανάμεσα στου Προέδρου των Επιτροπών του δύο Κοινοβουλίων. Αυτό θα διευκολύνει τι διμερεί σχέσει και έτσι τα δύο θεσμικά όργανα θα μπορέσουν να επιτείνουν τη συνεργασία τους. Ε, ξέρετε ότι πέρυσι ήδη ε, ε, έχουμε κάνει πάρα πολλές επισκέψεις επιτόπου στην Ουκρανία. Σας έχω επισκεφτεί και εγώ πολλές φορές και μπορείτε να δείτε την ανταπόκριση που δείχνουν οι συνάδελφοί μας διότι θέλουν να μετάσχουν σε αυτήν την διαδικασία. Επίσης, εσείς θα αποφασίσετε το δικό μου ε, το κοινοβούλιο που είναι πολύ μικρότερο από τη Ουκρανία έχει 28-29 επιτροπές. Μπορείτε να έχετε 28, μπορείτε, όπως εδώ στο κοινοβούλιο μπορεί να έχετε 20... Ε, εσείς θα το αποφασίσετε αυτό και ε, στο Κίεβο και στις Βρυξέλλες στους επόμενους μήνες ε, μπορούμε να δούμε πώς ακριβώς στην πράξη θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για τις επιτροπές. Για τον κύκλο του προϋπολογισμού τώρα. Ακούσατε κάποια, κάποιες σε κλειδιά εδώ στο Κοινοβούλιο που σε καθημερινή βάση ασχολούνται με τα βασικότερα νομοθετήματα που εγκρίνει το Κοινοβούλιο και με μία από τις βασικότερες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου είναι η έγκριση του προϋπολογισμού της Ένωσης και είναι πάρα πολύ στενά τα χρονοδιαγράμματα, είναι εξαιρετικά διαρθρωμένη διαδικασία και η εμπειρία μας μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο το Ουκρανικό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια διότι μπορείτε έτσι να προετοιμαστείτε για, όλα τις, για όλες τις υπόλοιπες πτυχές ε, της δουλειάς σας για την ευθυγράμμιση της χώρας σας ε, με τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω πέρα από τις δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει βάσει τη Συμφωνία Σύνδεσης. Και Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσετε το ρόλο που έχουν κάποιοι συγκεκριμένοι βουλευτές που έχουν ρόλο κλειδί ως προς τα θέματα του προϋπολογισμού για την διαφάνεια και τη λογοδοσία και τον αντιπροσωπευτικό ε, το, το ρόλο εκπροσώπησης ε, του, του, του Κοινοβουλίου. Εδώ μπορούμε να ανταλλάξουμε πρακτικές ε, και σας παραπέμπω εδώ στο, στη συμφωνία μεταξύ Σλισλίνσκι και ε, Βέλε για τη διοικητική συνεργασία των κοινοβουλίων, ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων, καλύτερη διαφάνεια ως προς τις εργασίες, επικοινωνιακή πολιτική του Ουκρανικού Κοινοβουλίου. Όλες αυτές οι διαστάσεις ε, μπορούν να ενισχυθούν με συγκεκριμένες προτάσεις που ακούσατε από τους γενικούς μας διευθυντές ε, εχθές ε, που, σας, ε, που εισηγήθηκαν τρόπους, πρακτικούς τρόπους ε, για να εφαρμοστούν αυτές οι συστάσεις. Επικοινωνία με τους πολίτες επίσης. Δύο χρόνια μετά το Μαϊντάν και γνωρίζοντας ότι οι μισοί βουλευτές είναι νέοι, προέκυψαν από την κίνηση από κάτω προς τα πάνω από τη βάση ε, και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι σημαντικό να ε, διαρθρώσουμε τη συζήτηση γύρω από την αρχή της συμμετοχικής ε, δημοκρατίας. Και χθες εμείς το απόγευμα κάναμε άλλη μια επικοινωνία, άλλη μια συζήτηση με συμμετοχή και από την Ουκρανική αντιπροσωπεία με δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται και εκεί και κάθε φορά που πηγαίνουμε κοιτάμε να δούμε τι κάνουν οι εκπρόσωποι τη Κοινωνία των πολιτών, των συνδικάτων και άλλων φορέων της κοινωνίας για την υλοποίηση της συμφωνίας. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια για το άνοιγμα, για τη διαφάνεια είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Συγκεκριμένα. Υπάρχει ιδέα να δοθούν απαντήσεις συγκεκριμένε ανταπόκριση καλύτερα σε συγκεκριμένα αιτήματα των πολιτών. Σε αυτό μπορεί η Επιτροπή των Αναφορών να το αναλάβει. Η Επιτροπή των Αναφορών δηλαδή η οποία επεξεργάζεται συγκεκριμένα αιτήματα και προσφύγια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάρη σε αυτήν δίνει με την ε, δέουσα διαδικασία το Κοινοβούλιο απαντήσεις στα αιτήματα και άρα μπορείτε να το υιοθετήσετε κι εσεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και βέλτιστες πρακτικές. Άλλο ένα θέμα που απασχόλησε πάνελ εργασίας εχθές. Είχα την ευκαιρία και εγώ μας με τον Όστοπ να ε, συμπροεδρεύσουμε δύο χώρες που κατά την θεώρησή μου είναι από τις πιο σημαντικές για την ε, Ουκρανία στην προσπάθειά της να διαγράψει αυτό το σημαντικό οδικό χάρτη. Το κεκτημένο λοιπόν, το οποίο συμπεριλαμβάνει πρωτογενή και και παράγωγη νομοθεσία, δικαστική πρακτική όπως αυτή έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 60 χρόνια και περισσότερο με πολύ απαιτητικές προδιαγραφές. Είναι δύσκολο δηλαδή να εισαχθεί το επίπεδο αυτό, αλλά υπάρχουν χώρε που έχουν καταφέρει να φτάσουν στο επιδιωκόμενο επίπεδο. Ο κύριο Αρουσβόλσκι μα περιέγραψε, μας με τον κύριο, με τον ε, πρέσβη μα περιέγραψαν την εμπειρία τη Πολωνία, που είναι πολύ σημαντική και λόγω τη γεωγραφική εγκύτητα και τη ομοιότητα. Άρα μπορεί σημείο αναφορά για εσά να είναι η Πολωνία. Ο κύριο Αντρόκοβιτ, υπουργό των εξωτερικών, τον εγώ ήμουν αντίστοιχα αρμόδιος για την διαπραγμάτευση εκ μέρους Κροατίας για, ε, για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και ε, εξελίξεις. Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά σε συνεργασία με όλα τα πλεκόμενα Υπουργεία, με κοινοβουλευτικό έλεγχο, πολύ δαπανηρή προσπάθεια άνευ προηγουμένου προσπάθεια μετάφρασης των 130.000 σελίδων της νομοθεσίας, γιατί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, για να μεταφραστεί σε μια γλώσσα σημαίνει και πολύ συστηματική δουλειά ενός διοικητικού μηχανισμού κρατικού, αλλά και ταυτόχρονα πολύ προσεκτική καθοδήγηση από τα ευρωπαϊκά όργανα και προσεκτική καθοδήγηση, θέλω να τονίσω αυτό, γιατί μερικές φορές το να στηρίζεται ε, κανείς μόνο στην, ε, μια, σε μια γενική και φυρημένα ιδέα του τι μπορεί να υπάρχει σε βάση δεδομένων και στο ίντερνετ δεν μπορεί να είναι αρκετό. Πολλές φορές δεν υπάρχουν πια τα έγγραφα τα οποία κανείς σκέφτεται να μεταφράσει και άρα χρειάζεται μεγάλη υποστήριξη και από τις μεταφραστικές μονάδες του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, του Συμβουλίου, του Δικαστηρίου, των Τραπεζών που είναι απαραίτητο να γίνει εγκαίρος και εφέτος αυτή η επικοινωνία μεταξύ των ε, αρχών των μεταφραστικών και των αντίστοιχων ουκρανικών υπηρεσιών μετάφρασης. Με την εναρμόνιση λοιπόν. Στην εναρμόνιση το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε δύο πτυχές. Πρώτον, να μην μετατραπείτε μόνο σε μια ε, σε μια σφραγίδα που θα δίνει την έγκριση. Δηλαδή να ενισχύσετε τη θεσμική σας δυνατότητα και ικανότητα ως προς την πραγματογνωμοσύνη σας. Δηλαδή το προσωπικό της ράντα να ενισχυθεί ως προς τις γνώσεις, να είναι πιο ε, πλούσιο το γνωστικό περιεχόμενο που έχουν να προσφέρουν και οι δικηγόροι που θα έχετε βεβαίω συνομικοί, αλλά και το λοιπό προσωπικό, ώστε να ελέγχεται και η σταγματικότητα των προτινομένων διατάξεων σε σχέση με το Εθνικό Σύνταγμα και βέβαια σε σχέση με το κεκτημένο η συμβατότητα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με μια διαδικασία πολύ σημαντική, πολύ κρίσιμη, είναι απαραίτητο να μην ε, υποκύψετε ενώπιον ε, ενός νομοθετικού τσουνάμι που σας περιμένει. Εγώ στη χώρα μου είχα να κάνω με 718 ε, παράγωγα και ε, πρωτογενή μάλλον κείμενα και 170 δευτερογενή ε, παράγωγα που έπρεπε να εισαχθούν στην νομοθεσία μας. Είναι λοιπόν τεράστιος όγκος αυτός ο νομοθετικός. Και ιδιαίτερα εδώ οι συνάδελφοι και από την ε, από το Κοινοβούλιο γενικότερα αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ε, ΡΑΝΤΑ μπορούν να αναλάβουν αυτό το δύσκολο και σημαντικό έργο. Επίσης, συμφωνούμε και καταλήγουμε ότι στις εξεμενιέ συναντήσει που θα έχουμε θα εξετάζουμε λεπτομερώς πολιτικές προτεραιότητες τη διαδικασία τη μεταρρύθμιση. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, την εναρμόνιση νομοθεσία. Κάθε φορά που θα συναντιόμαστε σε ένα επίσημο πλαίσιο, θα καταγράφουμε την πρόοδο αυτή τη διαδικασία εναρμόνιση για το ρόλο του Κοινοβουλίου και των πολιτικών κομμάτων, για τον ρόλο τη κουλτούρα, τη νοοτροπία, τη εξέβρεση συνενέσεων. Πρέπει νομίζω να κάνουμε τακτικές επαφές με το Ουκρανικό Κοινοβούλιο για να εμβλήσουμε το πρόβλημα πάνω απ' όλα πρέπει να ενισχυθεί ο διακομματικός διάλογος, να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας με τα αδελφά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να χτίσετε πάνω στις διαδικασίες που έχουν ε, αποδειχθεί σωστές με τη βοήθεια των όσων είπε και ο Πρόεδρος ε, Κόξ στα σημεία δηλαδή στα οποία δεν έχετε μεταξύ αποκλήσεις, στα σημεία στα οποία μοιάζεται και σε αυτό μπορεί να ενισχυθεί ο διακομματικός διάλογος και η επικοινωνία μεταξύ των κομμάτων. Και δύο-τρει γραμμέ μόνο για να καταλήξω στα συμπεράσματα. Ο πρόεδρο Κόξ ε, σημείωσε την ε, διάθεση του να προσφέρει και την διαθεσιμότητά του να προσφέρει βοήθεια σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ ευγενική χειρονομία Ξέρουμε πολύ καλά το ενδιαφέρον και τι στενέ σχέσει που έχει με τους Ουκρανούς συναδέλφου. Θα βρούμε λοιπόν κατάλληλες δομέ μα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να σα επιτρέπουμε και εσά να παρακολουθείτε τις ε, ε, να συμμετέχετε και να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες μας. Ίσως ε, όταν βρούμε μια ημερομηνία που θα σας ε, εξυπηρετεί και εσάς κύριε Κόξ και εμένα μπορούμε να πηγαίνουμε στο Κίεβο να παρακολουθούμε, να συναντούμε και να συζητούμε με τους συναδέλφους μας και βέβαια και με τη νέα αυτή συμφωνία διοικητική συνεργασίας μπορούμε να έχουμε ένα ρεαλιστικό οδικό χάρτη με τη συμφωνία και του Πρόεδρου Γκρόισμαν που θα ορίζει και τι συγκεκριμένε δραστηριότητε όπω θα πρέπει αυτέ να αναπτυχθούν. Επίση. και για να ολοκληρώσω πάνω σε ορισμένε πολιτικέ στοιχείε, γιατί στη τελευταία ανάλυση περί πολιτική διαδικασία πρόκειται. Έχουμε ένα πλαίσιο ανάπτυξη δυναμικού και δυνατοτήτων, αλλά εγώ έχω εντοπίσει τέσσερα κύρια σημεία. Πρώτον, ε, διαπιστώνω σημαντικό βαθμό πολιτικής οριμότητας που ξεφράσανε οι συνάδελφοι εδώ βούληση για διατήρηση της διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, ε, αίτημα υποστήριξης προς την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τα Εθνικά Κοινοβούλια, στην προσπάθεια αυτή και συγκεκριμένα ωφέλη. Διάγνωση συγκεκριμένων ωφελών και νομίζω ότι σε αυτό ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μερικέ παραπάνω λεπτομέρειε που θα πρέπει εσεί από πλευρά σα να υλοποιήσετε στι επόμενε εβδομάδε και έλαφρα προσπάθεια της Επιτροπής για μια επίσημη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου εσείς να ε, μπείτε στον κατάλογο των ε, κρατών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση του διαβατηρίου στις προσεχείς προτάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι και οι Ουκρανοί αν καταλάβουν ότι η Ευρώπη ε, δεν τους γεννά, δεν τους θέτει διοικητικά εμπόδια, γραφειοκρατικά εμπόδια, θα προχωρήσουν ακόμη περισσότερο. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το βελτιώσουμε πολύ στα επόμενα ένα-δύο χρόνια. Αυτέ λοιπόν τι λίγε προποθέσει θα πρέπει να υλοποιήσετε ακόμη. Επίση και εμεί πρέπει με την ε, καθοδήγηση των Γερμανών και Γάλλων ε, φίλων και στην υλοποίηση της συμφωνίας του Μίνσκ ε, να προχωρήσουμε αλλά και ιδιαίτερα να βοηθήσουμε σε ένα ειρήνα για την ειρηνική ε, επανένταξη των κατεχομένων αυτή τη στιγμή εδαφών με βάση τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξασφάλιση ειρήνης, συμφιλίωση μετά τη σύγκρουση, αμνηστία, ανοικοδόμηση, οργανώση ενωτευτών εκλογών, έλεγχο των συνόρων, συνεργασία με τους εταίρους και πα, διπλωματικές διευκολύνσεις, ώσπου, ώστε και πάλι να επαναταχθεί και πάλι αυτό το κομμάτι της επικράτειάς σας στη σταγματική σας τάξη. Δύο στρατηγική σημασία θέματα. Και αναφέρομαι όχι μόνο στον Τόνιας και το Λούγκαν, που είναι βέβαια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουμε εντοπίσει και τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν χάρη στη δουλειά και της ε, Επιτροπή κοινοβουλευτική συνεργασία. αλλά επίση και νομίζω ότι αυτό θα είναι από τα κύρια μηνύματα, Όλη τη ε, ιεραρχική δομή και των δομών του Κοινοβουλίου γενικότερα. Επίση πρέπει να σα πω ότι το Κοινοβούλιο ποτέ δεν είχε τέτοιου είδου και επίπεδου συνεργασία με άλλο κοινοβούλιο άλλη χώρα. Αυτό είναι πρώτη φορά στην ιστορία που συμβαίνει και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι και για μας αυτό το εγχείρημα το ευρωπαϊκό στο οποίο έχετε αποδηθεί. Δεν μπορούμε παρά να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους και εμείς από πλευράς μας συμβάλλοντας όσο μπορούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Ε, thank you, ε, thank you, Mr. for... Σας ευχαριστώ και εγώ για τις λεπτομέρειες με τις οποίες ε, στις οποίες αναφέρθηκες και που τόσο στενά συνδέονται και με τις συστάσεις. Με χαρά θα δώσω τώρα το λόγο στον Όψετ Τζίνιβαρ που είναι ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας ε, της Επιτροπής Σύνδεσης της Ράντα. Ε, θα ήθελα όμως αν μου επιτρέπετε πρόεδρε εγώ να μιλήσω ε, ουκρανικά.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 Αυτή η εκδήλωση που διαρκεί εδώ και ε, μια εβδομάδα στις Βρυξέλλες είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα ήθελα μάλιστα να σας ευχαριστήσω ε, τόσο τον πρόεδρο του Ισράντα όσο και τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον Μάρτιν Σούλτσε, για αυτή την πρωτοβουλία να ξεκινήσει ένα μια τέτοια εκδήλωση είναι εξαιρετικά σημαντικό χωρίς υπερβολή για το μέλλον του κοινοβουλευτισμού στην Ουκρανία και για τη μεταρρύθμιση της κοινωνίας ε, καθώ και για την αποδοχή από πλευρά τη επικοινωνία των πολιτών των μεταρρυθμίσεων αυτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο Πατ Κόξ για όλη τη δουλειά που έκανε ο ίδιο, ε, και οποία κράτησε αρκετές, ε, αρκετούς μήνες Ε, και αυτό δεν ήταν απλό. Ε, μπόρεσε να μας καλέσει, μπορέσαμε να εμπλακούμε στην προετοιμασία αυτής της ε, βαθύτατης ενδελεχούς και όρεμης έκθεσης. Η έκθεση αυτή δεν περιλαμβάνει οδηγίες, δεν περιλαμβάνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε. Μας δίνει μόνο τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε στην κατάσταση να καταγράψουμε, να βρούμε και να λάβουμε αποφάσεις, να βρούμε λύσεις και να λάβουμε αποφάσεις εμείς οι Και η συζήτηση, τα όσα είπε, ανέφερε και ο συνάδελφος Πλένκοβιτς, δικαιολογεί, αιτιολογεί μάλλον το ότι είμαστε έτοιμοι για μια τέτοια εργασία αυτομεταρρύθμισης και είμαι ευτυχής που Είναι προτεραιότητα η μεταρρύθμιση της Ουκρανικής ε, νομοθεσίας Δυστυχώς δεν είναι, δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ελπίζω πως θα καταφέρουμε να το καταστήσουμε πρώτη προτεραιότητα γιατί θυμόμαστε ότι ολόκληρη η προσπάθεια για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη δυνατή ε, μέσω της έκφρασης της βούλησης του λαού που φάνηκε στο Μαϊντάν και οφείλεται σε όλες αυτές τις ζωές που χάθηκαν. Αυτό δεν μας επιτρέπει να ξεχάσουμε δεν μας επιτρέπει να ξεχάσουμε ότι έχουμε τώρα την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια νέα χώρα και καλό όλους μας τους ε, εταίρους ώστε να επιταχύνουν και να κατανοήσουν ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε λάθος και να χάσουμε, να ιτηθούμε. Πρέπει να νικήσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης ε, γιατί τώρα που είμαστε κάπου στα μέσα γιατί έχουμε κάνει την ανάλυση, έχουμε συζητήσει την έκθεση όμως ε, δεν έχουμε ένα πλάνο δράσης, δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένα βήματα που να πρέπει να ακολουθήσουμε. Ελπίζω πως το Ευρωκοινοβούλιο και η αποστολή του Ευρωκοινοβουλίου ε, θα συνεχιστεί το καθήκον τι μας ε, θα είναι κάπως διαφορετικό και με ευτυχής που ο Πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία να να συνεχίσει την εργασία του στην Ουκρανία και εμείς στηρίζουμε βεβαίως αυτήν την θέση. Νομίζω πως η εντολή της Επιτροπής θα πρέπει να συνεχιστεί με κάπως διαφορετικά καθήκοντα. Αυτά είναι ήδη στην ημερήσια διάταξη και θα ήθελα να μπορέσουμε να το συζητήσουμε μαζί με τον συνάδελφο Πλένκοβιτς ε, για την εκτεταμένη ε, συνεδρίαση, ε, την συνεδρίαση του Διευρυμένου Προεδρείου της ε, Επιτροπής Συνεργασίας και Σύνδεσης. Μέσα σε αυτές τις αλλαγές που θα θέλαμε να υπάρξουν στο Κοινοβούλιο λοιπόν είναι και αυτή και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσω για την ε, θερμή και ομαλή εξέλιξη αυτή εδώ τη εκδήλωση. Ελπίζω ότι την επόμενη φορά δεν θα μιλήσουμε για το τι πρέπει να γίνει, αλλά θα, θα γιορτάσουμε για την επιτυχία του νέου μας κοινοβουλίου. Και θα βλέπουμε τα παλιά μόνο ως ε, ένα σημείο στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Σάμερεκ και σας ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή στην, ε, ε, που κάνατε στην εργασία αξιολόγησης, γιατί πολλές πόρτες ε, στο Κίεβο, άνοιξαν για μας. Εκτιμώ πολύ την δουλειά σας. Και τώρα με χαρά θα στραφώ στον Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Γραμματείς, και να τους καλέσω να υπογράψουν το έγγραφο που έχει να κάνει με την ε, δημιουργία και την οικοδόμηση διοικητικών υποδομών. Αυτή την εταιρική σχέση θεωρώ ότι είναι μεγάλο προνόμιο που βρίσκομαι σήμερα εδώ. για να είμαι παρόν σε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ πριν δηλαδή το κοινοβούλιο να γαλιάσει και να τόσο πολύ ένα άλλο κοινοβούλιο. Και αν υπάρχει ένα κοινοβούλιο σε ολόκληρο τον κόσμο που συμβολικά αυτό είναι πραγματικά ε, σημαντικό, είναι η σχέση με την Ράντα. Δεν, θέλω, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι, ή βέβαια ευχαρίστω αν το επιθυμείτε. Ίσως ο Κλάους και μετά ο κύριος Τιζίτσκι και μετά θα ε, υπογράψουμε το έγγραφο. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Πατ Κόξ. Είναι συναρπαστική η στιγμή, όχι μόνο για την εκδήλωση αυτή, αλλά γιατί είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει. Όπως εξήγησες, δεν έχει ξαναγίνει αυτό στο παρελθόν με οποιοδήποτε κοινοβούλιο. Πέραν αυτού όμως, Θυμάμαι στη Μαϊντάν να κυματίζει κεντρικά η ευρωπαϊκή σημαία και αυτό δεν είναι απόδειξη μόνο της βούλησης Ουκρανίας ε, να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σημαντική ενθάρρυνση για μας ε, διότι ορισμένες φορές ε, λόγω των προβλημάτων και των λεπτομεριών χανόμαστε λίγο, χάνουμε την γενική άποψη της κατάστασης και βλέποντας σε μια γειτονική χώρα να κυματίζει η σημαία μας, ε, μας θυμίζει ε, ποιος είναι ο στόχος μας. Υποστήριξη λοιπόν για τον εκδημοκρατισμό εχθές με τους γενικούς διευθυντές ε, του Κοινοβουλίου, με υποφαινόμενο αλλά και τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα συζητήσαμε και εστιάσαμε την προσοχή μας σε βασικά ζητήματα όπως ε, επιστημονική τεκμηρίωση, επικοινωνιακή, πολιτική, πληροφορική για να μην το ξεχνάμε και αυτό και τώρα αυτή η πολύ καλή συζήτηση θα μετατραπεί σε μια ε, ε, μακρά, μακροχρόνια, σταθερή και καρποφόρα διοικητική συνεργασία. Σας ευχαριστούμε κύριε Βέλε, ο κύριος Ξυζίνσκι. Ευχαριστούμε πρόεδρε Κόξ, Βλαντιμίρη Μπαρίσοβιτσε, κύριε Κλένκοβιτς, κύριε Βέλε. Θέλω να εκφράσω τη χαρά και την τιμή που νιώθουμε με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που έγινε κύριε Κόξ, διότι για μας, για την Ουκρανία, είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η συνεργασία, η ανάλυση που έγινε και ο εντοπισμός των προβλημάτων που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας μας δείχνει τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλουμε. Δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοια διοικητική συνεργασίας και για να εφαρμόσουμε το σχέδιο δράσης και τις συστάσεις θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Θα μεριμνήσουμε ώστε να στεφθεί με επιτυχία αυτή η συνεργασία και η γραμματεία του Κοινοβουλίου θα επιληφθεί όλων αυτών των ζητημάτων. Φυσικά υπολείπονται και άλλα πολλά προς συζήτηση. Έχουμε παρόλα αυτά ήδη αρχίσει πριν την υπογραφή της συμφωνίας την εφαρμογή αυτών των συστάσεων και θα θέλαμε να εκφράσουμε γι' αυτό την ευγνωμοσύνη μας προς τον κύριο Βέλλα. Ας ε, προβούμε λοιπόν στην υπογραφή της συμφωνίας. Hold up the, the, the signed documents there. Να κρατήσουμε ψηλά το έγγραφο όπως το υπογράψατε. Ας πούμε ότι είστε και εσείς αιρετοί πολιτικοί. Μην τρέψετε τις κάμερες. Σας ευχαριστούμε. Με χαρά λοιπόν τώρα απευθύνομαι στον κύριο Γκρόισμαν για να κλείσει τις σημερινές εργασίες. Και πρέπει να πω ότι με ενέπνευσαν ε, τα λόγια του Κλάου Βέλε για την ευρωπαϊκή σημαία που βρίσκεται πίσω μας. Το 2003, όταν είχα την τιμή να προεδρεύω του σώματος, προσεκλήθη σε μια εκδήλωση στην Αθήνα για να μιλήσω στην εκδήλωση υπογραφής των συνθήκων προσχώρησης των 10 τότε κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, Ευρωπαϊκή, Ελληνική Προεδρία, εν τη σοφία της, προσκάλεσε τον κάθε ηγέτη από κάθε ένα από τα 10 κράτη-μέλη και τον κάθε ηγέτη από τα 15 παλαιότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κάθε πρόεδρο Ευρωπαϊκού Οργάνου να λάβουν το λόγο. 28 το όλων ομιλητές, όπως καταλαβαίνετε ήταν βαρύ το πρόγραμμα και κοπιαστικό. Μετράγαμε 28, 27, 26, πόσοι μείνανε. Εγώ ήμουν από τους τελευταίους που έπρεπε να μιλήσουν στο τέλος εκείνης της ημέρας και έλεγα τι μπορώ να πω εγώ τώρα πια, όντας ο 27ος ή 28ος ομιλητής, μέσα σε τρία λεπτά. Και ευτυχώς περισσότεροι από τους ομιλητές και τους, συμβούλου, ε, συμβούλους και τους ερευνητές που είχαμε νωρίτερα ακούσει, είχαν μιλήσει για την αρχαία Ελλάδα, για τη δημοκρατία, για το λίκνο του πολιτισμού και όλα αυτά. Και, και έλεγα εγώ τώρα τι να τους πω εγώ που να αναφέρεται και στον ενωπιό χαρακτήρα της Ένωσης. Οπότε ζήτησα από τους ε, ε, συμβούλους μου να ψάξουν γρήγορα γρήγορα ποιο είναι το νόημα της ευρωπαϊκής σημαίας και από πού απορρέει. Λοιπόν, ήταν μια σημαία που υιοθέτησε το Συμβούλιο, του Ευρωπα... το Συμβούλιο της Ευρώπης στη δεκαετία του 50, όπου ζήτησαν από ειδικού σημεολόγους και συμβολολόγους να τους προτείνουν μια σειρά από σχέδια για σημαίες και ανακάλυψα με μεγάλη μου χαρά ότι αυτό το σχέδιο το είχαν ε, υποβάλει από την Ιρλανδία ένας δόκτωρ Σλέβεν, ε, ειδικό σε σύμβολα και οικόσημα της Ιρλανδίας. Με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν το διαπίστωσα αυτό εκείνη την ώρα. Αυτό το μπλε της σημαίας ήταν σύμβολο για τον ουρανό στη Βόρεια Ευρώπη. Βέβαια βρισκόμαστε στο Βόρειο ημισφαίριο. Ο κύκλος, ο σύμβολος σε οικόσημα, συμβολίζει την αρμονία. Το αστέρι είναι ένα σύμβολο το οποίο μας καλεί στην κοινή μας ε, μυθολογία και στις κοινές μυθολογικές βάσεις να κοιτάμε πιο μακριά, να μην κοιτάμε το καθημερινό και τη ρουτίνα. Το 12, ο αριθμός των αστεριών, για την εναλλαγή των μηνών και την εξέλιξη που πρέπει κανείς να παρακολουθεί όλα αυτά. Ο κύκλος λοιπόν των αστεριών δεν είναι κλειστός, είναι ανοιχτός σε όλους εκείνους οι οποίοι προσβλέπουν, οραματίζονται να μπουν μέσα στον κύκλο αυτόν. Μεγάλος ο συμβολισμός λοιπόν και είναι καλό να αναλογιζόμαστε τι σημασία έχει κάθε φορά που τα μετρήσουμε αυτή και όταν κάνουμε ό,τι κάνουμε αυτή την εποχή. Ευχαριστώ πολύ τους αδέλφους Πλάνκοβιτς και λοιπούς από την ε, ομάδα παρατηρητών των εκλογών. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο Σούλτς που ανέλαβε την ε, ηγετική αυτή δράση καθώς και τον πρόεδρο Κρόισμαν στην προσπάθεια για την ανοικοδόμηση συνενέσεων και βέβαια οπωσδήποτε την ίδια τη Βερχόβνα Ράντα. Το έγγραφο έχει το εξής ισχυρό σημείο ότι δεν ανήκει σε κανέναν και άρα ανήκει στους πάντες. Αυτό δείχνει μια ενότητα σκοπού που εκφράζεται εδώ στις Βρυξέλλες αλλά θα εκδηλωθεί και στο Κίεβο. Ο ρόλος της αποστολής της ίδιας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ένας εξωτερικός μεν μικρός δε χημικός καταλήτης αυτής της χημίας της συνενέσεως για την ίδια την Ουκρανία. Και για να κλείσω όπως ξεκίνησα και τις προάλλες παραθέτοντας τα λόγια του Ζώμονη του Μεγάλου Ιδρυτή ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς ανθρώπους και τίποτα δεν διαρκεί χωρίς θεσμούς. Μα προφανώς, αν δεν είχαμε μεγάλους ηγέτες ως άτομα που θέλησαν να δώσουν αυτή την εξέλιξη, δεν θα είχε ξεκινήσει τίποτα. Αλλά και δεν θα είχε μπορέσει να μετατραπεί σε μια θεσμική μορφή και να αναπτυχθεί. Και κλείνοντας λοιπόν, και παραδίδοντας το μικρόφωνο για αυτή την τόσο σημαντική εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στην Ουκρανία, θέλω προσωπικώς να αποτίσω θερμότατο φόρο τιμής στον εξεβονίμων κύριο, τον κύριο Γκρόισμαν, γιατί με τη δική του ηγεσία τη βούληση του να καθοδηγήσει, να ανοίξει πόρτες, πόρτες να είναι ανοιχτή σε όλους οι Βερχόβνα Ράντα, το πνεύμα αυτό του ανοίγματο και της ειλικρίνειας του πριστή είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε σε όλο τον κόσμο άλλωστε. Και νομίζω ότι έτσι δείχνεται και πόσο μεγάλη βούληση θέλετε, με πόσο μεγάλη βούληση θέλετε να προχωρήσετε στη μεταμόρφωση. Και ιδιαίτερα θέλω να τονίσω ότι δεν ζήτησε, δεν επεδίωξε η μεταρρύθμιση αυτή να φέρει τη δική του σφραγίδα, να είναι δική του μεταρρύθμιση. Θέλησε να είναι ολονών η μεταρρύθμιση, να φέρει τη σφραγίδα όλων σα. και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί η ηγεσία δεν σημαίνει είναι δικό μου και το κάνω τι θέλω. Η ηγεσία σημαίνει ορίζω μα με του άλλου στόχου και του επιδιώκω μαζί με του άλλου. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα του κύριου Κρόισμαν και με μεγάλη χαρά τώρα τον καλό να κηρύξει το πέρας των εργασιών τη εβδομάδα της Ουκρανίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμε ε, Πρόεδρε κύριε Κόξ, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι εδώ σήμερα μαζί σας και να που συνεργάστηκα μαζί σας τις τελευταίες τρεις μέρες αλλά και παλιότερα ε, μπορέσαμε να συλλέξουμε πολύ εμπειρία η πρωτοβουλία για αυτήν την ε, πρωτοβουλία, την Ευρωπαϊκή ε, Εβδομάδα της Ουκρανίας στο Ευρωκοινοβούλιο, έδωσε τη δυνατότητα σε εμά και στους συναδέλφους από την Ουκρανία να οικοδομήσουμε διόδους επικοινωνίας που δεν υπήρχαν μέχρι χτες μόλις. Ε, σήμερα συνεννόμαστε πολύ καλύτερα, καταλαβαίνόμαστε πολύ καλύτερα, καταλαβαίνουμε τα, πώς έχουν τα πράγματα στην Ουκρανία και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την... να καταβάλουμε τις προσπάθειες που χρειάζεται Δεν θα πρέπει να μακρηγορήσω, αλλά θα πρέπει κανείς να λέει αυτό που αισθάνεται. Βέβαια η χώρα μας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα εκτός ε, μιλώ για την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα, αλλά αντιμετωπίζουμε και εσωτερικά προβλήματα, μιλώ για την οικονομία, για το δικαστικό σώμα, μιλώ για το σχηματισμό αποτελεσματικών μηχανισμών, για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Όλα αυτά απαιτούν ε, ενοποιημένη εικόνα για το τι πρέπει να κάνουμε και προθέσεις. Πρέπει λοιπόν να προτάξουμε τα όσα πρέπει να γίνουν, πρέπει να προβούμε σε αναλύσεις αλλά και σε μια διάγνωση ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να αλλάξουμε. Συχνά έχω τονίσει ότι ένα από τα κύρια προβλήματα στην Ουκρανία είναι η θεσμική αδυναμία της χώρας. Ότι δηλαδή οι θεσμοί, οι κυβερνητικοί δεν αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα. Ως έχει πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την ε, οικονομία μας πρέπει να βελτιώσουμε το δικαστικό μας σύστημα ώστε να μπορεί ο κόσμος να το πιστεύεται πλήρως. Πρέπει να ενημερώσουμε τη... και να μεταρρυθμίσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες, να αποκεντρώσουμε το κράτος, να αναπτύξουμε τη δημοκρατία. Όμως όλα αυτά, όλα τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμίσεων εξαρτώνται από τον επαγγελματισμό μας, τις ικανότητές μας. Μιλήσαμε για κάποιες μεταρρυθμίσεις που δεν ήταν επιτυχείς, όταν η κοινωνία δεν ε, αισθάνεται ότι έγιναν μεταρρυθμίσεις. Ε, ίσως θα πρέπει να θέσουμε και να ρωτήσουμε και το συμπολίτε μας. Αντιδρούμε σωστά, να διερωτηθούμε. Αντιδρούμε σωστά στις ανάγκες της κοινωνίας, αντιμετωπίζουμε σωστά τις κρίσεις που ε, εμφανίζονται. Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτές όλες τις προκλήσεις χρησιμοποιώντας παλιά συστήματα. Αυτή είναι η ουσία να βελτιώσουμε τον τρόπο λήψης αποφάσεων, να βελτιώσουμε την ποιότητά μας. Έχουμε εκτελεστικό, έχουμε δικαστικό σώμα, έχουμε νομοθετικό σώμα, αλλά πρέπει να αλλάξει το σύστημα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ επαγγελματικοί και επιμελής. Η συνεργασία μαζί σας, μαζί με τον κύριο Κόξ, με τον κύριο Πλένκοβιτς, αλλά και με τη βοήθεια του Πρόεδρου Σούλτς, η δουλειά που έχει ενώσει τους Ουκρανούς ε, βουλευτές, τους Ευρωβουλευτές, αυτή η εργασία θα πρέπει να γίνει σωστά το νομοθετικό σώμα να είναι αυτό όπου η μεταρρυθμιστική αναζωογόνηση της ίδιας της Ουκρανίας θα ξεκινήσει. Ε, το Κοινοβούλιο θα είναι αυτό το οποίο πρέπει να αντιδράσει σωστά στις προκλήσεις, να δείξει σε όλους πώς θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η χώρα, η δημοκρατία, να σχηματιστεί το εκτελεστικό της χώρας μας για δεκάδες χρόνια, δεκαετίες μάλλον. Δεν υπήρχε μεταρρύθμιση. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι κατάλληλος ο κρατικός μηχανισμός. Πρέπει να μεταρρυθμιστεί και το δικαστικό σώμα, αλλά να είναι πραγματικό αποτελεσματικό. Δεν έχουμε πλέον χρόνο να κάνουμε μεταρρυθμίσεις προς χάρη των μεταρρυθμίσεων. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει το ποιοτικό αποτέλεσμα. Μόνο τότε θα μπορέσει η Ουκρανία να είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Και το λέω αυτό διότι έχουμε ένα καλό σχέδιο, αλλά πρέπει και να εφαρμοστεί σωστά. Χρειάζεται λοιπόν κοινό σχέδιο, πρόγραμμα δράσης και να δείξουμε υπευθυνότητα ώστε αυτό να το μετατρέψουμε σε πραγματικότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι κάθε αρχηγός κράτου, ε, κόμματος θα πρέπει να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων για το σύνολο της Ουκρανικής κοινωνίας. Δεν ανοίξαμε τις πόρτες, ανοίξαμε τις καρδιές μας εδώ, ανοίξαμε τις καρδιές μας στην Ευρώπη και θα θέλαμε αυτό να το ε, Μιλάμε για το καθεστώς, για το σιδηρούν παραπέτασμα που πρέπει να πέσει. Δεν θα πρέπει πλέον να μας χωρίζει τίποτα ε, να μπορέσει έτσι η Ουκρανία να μπει στην οικογένεια την Ευρωπαϊκή. Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος θα πρέπει να είναι ε, ειρηνική και ελεύθερη. Χωρίς πόλεμο πια. Όχι όπως τώρα που αντιμετωπίζουμε τέτοια πολεμική σύρεξη στην Ουκρανία. Είναι τεράστια αυτή η πρόκληση το έχω τονίσει και δεν μπορώ παρά να το ξαναπώ ότι και κάποιος είπε ότι η Ουκρανία είναι κομμάτι της Ευρώπης, ο πρόεδρος Σούλτς το είπε. Όχι, ε, το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει κουραστεί από την Ουκρανία. Το μέγεθος των προκλήσεων απαιτεί να είμαστε ε, στεναροί Γι' αυτό και όλοι μας, όλοι οι βουλευτές του Ουκρανικού Κοινοβουλίου, όλοι μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε και να πούμε ότι εμείς η αποφασή μας θα καθορίσει το πώς θα είναι η Ουκρανία στο μέλλον. Πώς θα ληφθούν αυτές οι αποφάσεις γρήγορα, όπως σήμερα, τα τραπάτρα ή θα πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα, μια χώρα όπου όλοι θα είναι καλύτεροι ποιοτικά. Εγώ ε, νομίζω πως θα πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο της ε, θεσμικής ορθότητας, ε, της επαγγελματικής ανταγωνιστικότητας και να μπορέσουμε να υιοθετούμε τις πολύ απαραίτητες αποφάσεις. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Σούλτς, τον κύριο Πλένκοβιτς, εσάς πρόεδρε Κόξ που κάνατε τόσο σπουδαία δουλειά και μάλιστα ε, θα έλεγα ότι το θεωρήσατε ότι είναι η δουλειά σας και όχι μόνο, το πήρατε προσωπικά. Και τώρα με την βοήθεια της ευρωπαϊκής κοινότητας μπορούμε από κοινού να δούμε ε, πώς θα προχωρήσουμε από κοινού. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες επάρσεις, όχι. Πρέπει να ε, συνεδριάσουμε εκ νέου και να εφαρμόσουμε τα όσα πρέπει. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Σας καλώ να συνεργαστείτε όλοι μαζί και ελπίζω πως έτσι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το έργο που έχουμε ενώπιον μας είναι σημαντικό να το συζητάμε. Είναι μεγάλη παράδοση. Ε, νομίζω πως έτσι μόνο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ποιοτική ε, λήψη αποφάσεων. Ε, ευχαριστώ και είμαι βέβαιος ότι τα καταφέρουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίαση αυτή. Για όσους επιστρέφουν στην Ουκρανία απόψε, και εγώ θα είμαι στο ίδιο αεροπλάνο. Ε, ελπίζω και εύχομαι καλή, καλό ταξίδι. Σλάμπα η Ουκράινα, είπε ο πρόεδρος, μάλλον στα Ουκρανικά.